Καλησπέρα σας πάντα. Τις Δευτέρες ξεκινάμε μια μικρή καθυστέρηση της συνεδρίασή μας. Αλλά αυτά έχουν οι Δευτέρες. Οι περισσότεροι έρχονται τη Δευτέρα, οπότε φτάνουν οι πτήσεις τους αργά. Μια και πέρασα όμως σχεδόν το ακαδημαϊκό τέταρτο, ας ξεκινήσουμε. Σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη, το σημείο 9, την ενημέρωση ε, για την πορεία των τριμερών διαλόγων για τα βιολογικά προϊόντα, αναβάλλεται για την επόμενη μας συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, παρακαλώ να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Έχουμε απευθεία αναμετάδοση στο διαδίκτυο της συνεδρίασης. Α, αλλά επειδή η αίθουσα χρειάζεται στις υπηρεσίες για μια συνεδρίαση πολιτικής ομάδας 6.30, πρέπει να ολοκληρώσουμε λίγο πριν τις 6.30. Έχουμε λοιπόν και διερμηνία 21 γλώσσες με εξαίρεση στα μαλτέζικα και ιρλανδικά. Για το σημείο 4 έχει προβλεφθεί επιπλέον διερμηνία σλοβακική και τσεχική. Να εγκρίνουμε για τα πρακτικά της 15ης Μαΐου και 29ης 30ης Μαΐου κατά τη συνηθισμένη διαδικασία και να περάσουμε στο κυρίως θέμα το σημείο 4 και να καλωσορίσουμε ιδιαίτερη χαρά τρεις Υπουργούς Γεωργίας την κυρία Γκαμπριέλα Ματετσνά που είναι Υπουργός Γεωργίας της Σλοβακίας και μάλιστα είχαμε συναντηθεί με την Υπουργό στη διάρκεια της Σλοβαϊκής Προεδρίας. Ε, μας είναι οικία λοιπόν. Πολύ πετυχημένη και αξιόλογη η Σλοβαϊκή Προεδρία. Επίσης έχουμε μαζί μας τον Τσέχο Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Μαριάν Γιουρέτσκα, καθώς και τον Σλοβαίνο Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Ντέγιαν Ζίνταν. Τους ευχαριστώ θερμά και τους τρεις ε, και για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν και για την ε, σημερινή τους παρουσία. Ε, μάλιστα εξέδωσαν έναν επίσημο έγγραφο με θέμα τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, αντιμετώπιση αθέμητων εμπορικών πρακτικών και βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αυτή. Ε, μαζί με τη Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λετωνία, Λιθουανία, παρουσίασαν αυτό το ανεπίσημο έγγραφο στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλίας στις 6 Μαρτίου και έτυχαν υποστήριξη από την Πολωνία, Ελλάδα, Κροατία, Βέλγιο, Κύπρο και Ρουμανία. Σας έχουμε μοιράσει μάλιστα το σχετικό έγγραφο, το ανεπίσημο. Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό που πολύ συχνά μας έχει απασχολήσει σε πολλές περιπτώσεις και επ' ευκαιρία πολλών συζητήσεων. Έχουμε επιληφθεί επανειλημμένως λοιπόν αυτών των θεμάτων, των αθέμητων εμπορικών πρακτικών και της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα φοδιασμού τροφίμων. Και μάλιστα είχαμε και έκθεση για το θέμα αυτό. Ζητήσαμε από την Επιτροπή να αναλάβει δράση Ε, δεν χρειάζεται να σε εξηγήσω καν γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα. Θα μας το εξηγήσουν οι καλεσμένοι μας. Πάντως ε, είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το θέμα αυτό και μας είναι προσφυλές. Μάλιστα, πέρσι το φθινόπωρο απευθύναμε έκκληση στον Επίτροπο Χόγκαν να επιταχύνει τις εργασίες προκειμένου να θεσπιστούν και νομοθετικά μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Γιατί ναι, μεν ορισμένε χώρε έχουν εθνικέ διατάξει για το θέμα αυτό, για την αντιμετώπιση του, αλλά χρειαζόμαστε και πανευρωπαϊκό δίκαιο, ενωσιακό δίκαιο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, μια και έχουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν κοινέ ρυθμίσει και κοινέ λύσει που θα είναι πιο αποτελεσματικέ από τι μεμονωμένε εθνικέ διατάξεις. Φαντάζομαι για όλα αυτά θα μας μιλήσουν και οι κύριοι Ντεκάστρο και Ντες, γιατί στη, στην πρόταση αυτή περιλαμβάνονται και στον κανονισμό, οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται και στον κανονισμό Omnibus, για τον οποίο είναι συναρμόδιοι οι δύο συνάδελφοι. Θα δώσω όμως το λόγο στους καλεσμένους μας πρώτα και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Δεν θα σας περιορίσουμε στο χρόνο αγόρευσης, αλλά παρακαλώ δείξτε κάποια εγκράτεια στη χρήση του χρόνου. Παρακαλώ. Πρώτα η Υπουργός από τη Σλοβακία. Ε, καλησπέρα σε όλους και σε σένα, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριοι βουλευτές. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τη διοργάνωση αυτής της συζήτησης. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα οποία δείχνουν στήριξη στις διάφορες πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, το θέμα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών για τη Σλοβακία είναι από τα πιο λεπτά θέματα και από τις πιο μακροπρόθεσμες προτεραιότητές μας. Εκτιμούμε πάρα πολύ το ενδιαφέρον που δείχνει το Κοινοβούλιο, το και η Επιτροπή για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Πρόσφατα στην ε, διατροφική αλυσίδα έγιναν σημαντικές διαρθωτικές αλλαγές. Υπήρξε μια συγκέντρωση πολύ έντονη φορέων δηλαδή επιχειρήσεων κτλ. Και, και που λειτουργούν στον γεωργοδιατροφικό τομέα. Και καθώς έγινε αυτή η συγκέντρωση, οι αγρότες έγιναν πιο, ο πιο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι σε, θέμα, σε θέση να προασπιστούν τα συμφέροντά τους και δεν μπορούν να εισπράξουν τα απαραίτητα ούτε για να καλύψουν τα έξοδά τους. Έχουν γίνει διάφορες ε, καταγγελίες σε εθνικό επίπεδο που καταγγέλουν τις πρακτικές κάποιων σούπερ μάρκετ που εκμεταλλεύτηκαν την ε, δεσπόλουσα θέση τους. Ήδη από το 2012 στη Σλοβακία προτείναμε ένα εθνικό νόμο για τις ε, άνισες και άδικες ε, συνθήκες ή σχέσεις στο εμπορικό τομέα και κυρίως στο γεωργοδιατροφικό τομέα. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει νομίζω σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγο ή πολύ. Το θέμα συζητήθηκε πολλές φορές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο υπουργό μας εκτιμάει την δράση της Επιτροπής και η προσπάθεια της Επιτροπής είναι να προωθήσει κάποιες εθελοντικές πρωτοβουλίες για την τροφική αλυσίδα. Πρέπει όμως δυστυχώς να παρατηρήσουμε ότι παρότι οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία αυτή προσπαθούν να εξαλείψουν όλες τις μορφές αθέμητων εμπορικών πρακτικών, αυτή η λεγόμενη πρωτοβουλία στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Εδώ και πολύ καιρό, σε διάφορα επίπεδα, βλέπουμε την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρξει μια νομοθεσία, μια κοινή νομοθεσία, ενωσιακή δηλαδή νομοθεσία. Αυτό το θέμα έγινε και μία από τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας μας πέρυσι στο Συμβούλιο. Η Προεδρία μας Έκανε προσπάθειες, ε, επιτυχής θεωρούμε και πιστεύουμε ότι μετά από πάρα πολλές πιέσεις, ε, μετά από πολλές εκκλήσεις, φτάσαμε σε επίπεδο συμπερασμάτων Υπουργών Γεωργίας και Αλίας. Δηλαδή φτάσαμε μέχρι να έχουμε συμπεράσματα σε αυτό το επίπεδο. Ε, επίσης προωθούνται ε, νομοθετικά μέτρα και μη νομοθετικά μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε στήριξη από όλου του υπουργού για αυτέ τι πρωτοβουλίε. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2016, επί Σλοβακικής Προεδρίας, καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Η Προεδρία μας δεν τελείωσε αυτή τη μάχη όμως. Το Μάρτιο του 2017 συμμετείχε σε μια πρωτοβουλία όπου συμμετείχαν διάφορες χώρες και που τον καρπό αυτής τη προσπάθεια σας τον παρουσιάσουμε σήμερα και θα είναι και η βάση για μια μελλοντική προσπάθεια προκειμένου να ενισχύσουμε τη θέση των γεωργών για να αντιμετωπίσουν τις αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές στο γεωργοδιατροφικό τομέα. Χαιρόμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα του φαινομένου και την επίπτωση που έχει στους γεωργούς και τη ζωή τους. Τώρα θα ήθελα να καλέσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν να προσπαθήσουν τόσο ώστε να υπάρξουν αποτελεσματικέ λύσει το συντομότερο δυνατόν, τόσο ώστε να μειωθεί η επίπτωση του προβλήματο αυτού. Είμαι πεπισμένη ότι από κοινού θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα και θα υπερασπιστούμε τον πιο αδύναμο κρίκο της γε... γεωργοδιατροφικής αλυσίδας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν το κυρίως θέμα, ή μάλλον ένα τα σημαντικότερα θέματα της Σλοβακικής Προεδρίας και το θέσατε ιδιαίτερα στην, στο Συμβουλίο Γεωργίας. Μάλιστα διοργανώσατε και μία σημαντική διάσκεψη με συμμετοχή πανεπιστημιακών κύκλων και εμπειρογνωμόνων. Ε, δώσατε ιδιαίτερα προσοχή στο ζήτημα αυτό. Όπως είπα, το θέσατε και στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλίας και περιλήφθηκε και στα συμπεράσματα της Προεδρίας. Σας ευχαριστούμε την κυρία Γκαμπρίελα Ματεσινά και δίνω το λόγο στον Τσέχο Υπουργό Γεωργίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την πρότασή μας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Βρισκόμαστε σε μία άνευ κατάσταση, γιατί έχουμε αυτή την πρωτοφανή περίπτωση να εμφανίζονται στην Επιτροπή Γεωργίας τρεις Υπουργοί Γεωργίας για να σας παρουσιάσω το θέμα αυτό, κάτι που μαρτυρεί την σπουδαιότητα που έχει για τα κράτη-μέλη. Μάλιστα συντάξαμε και έναν επίσημο έγγραφο για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το θέμα σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας. Όταν όμως ε, συζητούμε με τους ομολόγους μας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα γεωργοδιατροφικά προϊόντα γιατί διαπιστώνουμε ότι η θέση των γεωργών στην αλυσίδα, στην τροφική αλυσίδα είναι ένα κέριο ζήτημα, ένα θέμα θεμελιώδους σημασίας και μάλιστα ένας κοινός προβληματισμός των κρατών μελών. Οι αθέμετες εμπορικές πρακτικές είναι πρακτικές που ε, αποδεικνύουν την ανισορροπία που υπάρχει στις εμπορικές συναλλαγές σε αυτόν τον κλάδο. Και μάλιστα ε, προτείνουμε ισορροπημένους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με νομοθετικά μέτρα που θα ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε τομείς όπως ενέργεια, τηλεπικοινωνίες ή άλλους κλάδους όπου έχουμε διαπιστώσει ανισόρροπη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς λόγω της, του κατακαιρματισμού των διατάξεων. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τη μείζων αυτή πρόκληση, αντιμετώπιση αυτού του κατακαιρματισμού λόγω της ε, πληθώρας των εθνικών διατάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, είχαμε πρόσφατα το πρόβλημα της περιαγωγής και καταργήσαμε τα τέλη περιαγωγής. Είδαμε πόσο σημαντικά είναι τα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δεν είχαμε μια ευρωπαϊκή θέση και ένα ευρωπαϊκό μέτρο για τα τέλη περιαγωγής, δεν θα είχαμε επιτύχει το στόχο μας για την κατάργηση των τελών αυτών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλουμε λοιπόν να συμβάλλουμε και στο γεωργικό κλάδο στη βελτίωση της θέσης του γεωργού στην ε, τροφική αλυσίδα. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Πρόκειται για πρακτικές που ξεπερνούν το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και δεν αφορούν μόνο τα κράτη-μέλη και τους προμηθευτές τους, α, γιατί ακούμε μερικά επιχειρήματα που λένε ότι κάποιοι ε, πάροχοι υπηρεσιών και κάποιοι προμηθευτές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση κάτι που θέτει ένα αμφιβόλο και την ίδια του στην επιβίωση και λειτουργία. Επίσης, οι ρυθμιστικές αρχές, οι ελεκτικές αρχές δεν μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο τους γιατί δεν υπάρχουν αρκετά νομοθετικά μέτρα ή ρυθμίσεις που να επιτρέπουν ε, επαφή και ανταλλαγή απόψεων με άλλα κρατημέλη γιατί δεν έχουμε τέτοια πανευρωπαϊκά μέτρα. Γι' αυτό και οι Υπουργοί Γεωργίας, τα Υπουργεία Γεωργίας δεν έχουν αρκετούς μηχανισμούς ή εργαλεία ώστε να επικοινωνήσουμε τους ομολόγους τους και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες ενός ε, φορέα εκμετάλλευσης ή οικονομικού τελεστή και να κρίνουν κατά πόσο οι πρακτικές του είναι αθέμητες ή όχι. Επίσης, κάποια εθνικά νομοθετικά μέτρα δεν επαρκούν. Εξού και το πρόβλημα το οποίο επισημάναμε στο ανεπίσημο μας έγγραφο και που αφορά πολλές χώρες. Θέλουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να βρουν μια λύση. Είπατε κύριε Πρόεδρε πριν από λίγο ότι έχετε γύψει επανειλημμένως σε αυτό το θέμα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα. Απλώ εξετάζουμε, απλώς ε, συζητούμε για το θέμα αυτό. Γι' αυτό και συντάξαμε έναν επίσημο έγγραφο με τη διάγνωση του φαινομένου, την αναγνώριση της ύπαρξης των αθέμητων εμπορικών πρακτικών και που υποβάλλουμε κάποιες προτάσεις για το τι επιδιώκουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να δώσουμε μια νέα πνοή σε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί το 38% του κοινοτικού προϋπολογισμού ε, προορίζεται για την κοινή γεωργική πολιτική. Αρκεί όμως αυτή η πολιτική για να εξασφαλίσει την επιβίωση της γεωρικής δραστηριότητας των γεωργών μας, των αγροτών μας. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσαμε πολλοί άριθμες κρίσεις. Μπορέσαμε να τις αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, κρίση στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι τιμές γάλακτος έχουν καταβαραθρωθεί, έχουν μειωθεί πάνω από 30% ποια είναι η επιρροή αυτής της κατακόρυξης πτώσης ε, των ε, γαλακτοκομικών τιμών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους, στην καθημερινότητα των γιωργών. Προσπαθήσαμε με τον κοινοτικό προϋπολογισμό να βοηθήσουμε τους γιωργούς και τις οικογένειές τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αλλά και η κατάσταση δεν είναι ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη ή δεν είναι ίδια για όλους τους καλλιεργητές ή τους γεωργούς ή τους κτηνοτρόφους ή ε, όλους τους προμηθευτές. Βρίσκομαι ενώπιόν σας ως ε, υπουργό Γεωργίας, ως υπεύθυνο δηλαδή για εκατομμύρια οικογένειες ε, γεωργών και κτηνοτρόφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ήθελα η τροφική αλυσίδα να παρουσιάζει ανισορροπίε. Θα πρέπει κάθε κρίκο αυτή τη αλυσίδα, άρα και οι γεωργοί, να έχουν ε, ένα δίκαιο μερίδιο σε αυτή την αλυσίδα. Δυστυχώ, αυτή την ισορροπία τη τροφική αλυσίδα, διαταράσσουν και στρεβλώνουν οι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ και οδηγούν στη χρεοκοπία πολλού γεωργού. Ε, πολλοί αναγκάζονται να παράγουν σε τιμέ κάτω του κόστου η κατάσταση είναι αφόρητη και μη βιώσιμη. Θα πρέπει λοιπόν να μας βοηθήσετε να προετοιμάσουμε κάποιες νομοθετικές προτάσεις και να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτών των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα ο λόγος στο Σλοβαίνο Υπουργό Γεωργία, στον κύριο Ζίνταν Δέιαν. Παρακαλώ. κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, να καλωσορίσω και τους λοιπόν προσκεκλημένους. Ε, κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ καταρχάς ε, για το γεγονό ότι σήμερα καλέσατε εμάς τους τρεις ε, υπουργού σε αυτή τη σημαντική συνεδρία της Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου κάποιες προσθήκε να κάνω. Στην γεωργική παραγωγή, οι κρίσει ε, αποτελούν ε, μια μετάβλητη κατάσταση, γιατί όταν μειώνονται οι τιμές, δεν φορτώνεται ο γεργός ε, που δεν μπορεί να πουλήσει το γάλα του. Και πολύ απλά αναγκάζεται να αποδεχτεί ότι αυτό θα φορτωθεί την κρίση. Όταν βελτιώνεται η κατάσταση και αναπτύσσεται η οικονομία, η ανάπτυξη αυτή ουσιαστικά δεν φτάνει στη Γεωργία και έχουμε διαπιστώσει ότι το χάσμα μεταξύ του μικρού παραγωγού και των ε, τιμών των πρώτων είναι όλο και πιο μεγάλο και διαπιστώνουμε ότι είναι όλο και πιο πολλές οι κρίσεις που μαστίζουν τα... την οικονομία και όλο και λιγότερες απαντήσεις δίνονται στις κρίσεις αυτή στην ε, Σλοβενία υπογράφτηκε το 2011 ένας εθελούσιος κώδικας ε, συμπεριφορά και ο κώδικα, λοιπόν αυτός βελτίωσε κάπως ε, την κατάσταση. Κατέστησε την κατάσταση κάπως πιο διαφανή. Υπάρχουν ε, καθαρές ε, τιμέ πλέον που προβλέπονται. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες κακέ πρακτικές που έχουν παραμείνει, αλλά η κατάσταση γενικώ πως είναι πιο διαφανής και αυτό αποτελεί μια βελτίωση της κατάστασης και έτσι λοιπόν το 14 ψηφίσαμε μία μεταρρύθμιση του νόμου για τη γεωργία, όπου προβλέπεται και ένα άρθρο για την ε, διατροφική αλυσίδα και έτσι αναφέρονται και καταγγέλλονται οι λανθασμένες πρακτικές ε, στην αλυσίδα παραγωγή τροφίμων. Έχουμε θέσει ανώτατα ποσά για την προθεσμία πολυρωμής, 45 ημέρες κατά ανώτατο όριο. Και επίση δημιουργήθηκε και ένα διαμεσολαβητή για την τροφική ασφάλεια. Επίση ορίσαμε και κυρώσει και ο διαμεσολαβητή πλέον ε, υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια. Έχει βελτιώσει την κατάσταση, αλλά παρ' όλα αυτά η κατάσταση δεν είναι ακόμα η ευκταία. Η γεωργοί είναι ενωμένοι, αλλά όχι αρκετά. Και αυτό το βλέπουμε σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, υπάρχει ε, μια ένωση. Έχουμε και την βιομηχανικό, τον κλάδο της παραγωγής τροφίμων. Ίσως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει και κάποια αλληλεγγύη, αλλά δεν υπάρχει ισορροπία στις δυνάμεις και έτσι το 2004 διαπιστώσαμε ότι στην αλυσίδα διατροφική υπάρχουν πάρα πολλές ε, μετοχές στην παρούσα φάση πάρα πολλές προσφορές σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, πατάτε, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα τα οποία απολούνται και Νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην πέφτουν οι και επίσης θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στους αγρότες να παράγουν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βιώσιμη δουλειά Και επίσης θα πρέπει να επιλεχθούν αυτά και σε διεθνέ επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν και ε, συνήλθαμε με τους υπόλοιπους υπουργούς ε, Γεωργία. Θέλουμε λοιπόν να συμμετέχουμε για, την, ε, για κάποιες κατευθυντηρίες γραμμές προκειμένου να δοθεί ένα κοινό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί το πρόβλημα αυτό είναι ευρωπαϊκό. Πρέπει επίσης να ορίσουμε ποιες είναι οι αθέμητες πρακτικές. Ε. Επίσης προτείνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να οριστούν και κυρώσεις, ε, αν θέλουμε να καταγγείλουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ε για να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, συγκεκριμένε υπηρεσίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαμεσολαβητέ και άλλα τέτοια, άλλες τέτοιες υπηρεσίε. Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι ωφελούν και ότι κάθε κράτο πρέπει να λαμβάνει τι ευθύνε του. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, εδώ και κάποια χρόνια όλοι έχουμε αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει επαρκής ρύθμιση στη διατροφική αλυσίδα και ο πιο δυναμός κρίκος έχουμε διαπιστώσει ότι είναι ο γεωργός και επιτέλους θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην κατάσταση αυτή. Δεν μπορούμε να παραμένουμε απλά στην διαπίστωση των φαινομένων. Θα πρέπει τέλος να δράσουμε και ο επόμενο ο αρμόδιος επίτροπος θα έλθει αύριο στην Επιτροπή και τώρα λοιπόν πραγματικά αναμένουμε να συζητήσουμε πώς θα αντιδράσουμε, τι θα κάνουμε συγκεκριμένα και όχι απλά να παραμείνουμε στα σχέδια και στα πλάνα, προκειμένου να υπάρξει κάποια σωστή ανταπόκριση. Αγαπητοί ευρωβουλευτές, ε, θα ήθελα να σας ζητήσω να καταφέρουμε κάτι σημαντικό και συγκεκριμένο εδώ στην Επιτροπή σας για τους γεωργούς. Ευχαριστώ Δεκάστρο. grazie Presidente, grazie naturalmente ai σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερως για την ευκαιρία που έχουμε να ανταλλάξουμε ε, απόψεις με τρεις υπουργούς γεωργίας από κράτη-μέλη και να συζητήσουμε το θέμα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Μαζί με τον συνάδελφο Ντέσεν, μέρη και με τον κύριο Νταντέν, αλλά και με όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής, επεξεργαστήκαμε την έκθεση για τον κανονισμό Omnibus. Και στον κανονισμό Omnibus αδράξαμε την ευκαιρία και προτείναμε κάποιες ειδικέ διατάξεις με βάση το, την προεργασία που κάναμε στα πλαίσια και τις έκθεσης Μαγκίνες για το θέμα αυτό. Θα ήθελα, εν συντομία, να κάνω κάποιες, κάποιες μνήες. Για παράδειγμα, την υπεροχή των κανόνων της κοινή οργάνωσης αγοράς σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Αυτό είναι ένα κεντρικό σημείο του κανονισμού Omnibus, κάτι που αναφέρεται και στον επίσημο έγγραφό σας. Επίσης, υποχρεωτική γραπτή σύναψη συμβάσεων. Το είπαμε και στην Επιτροπή μας, το έχουμε συζητήσει ε, ευκαιρία και της προηγούμενης μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ρήτρα αναθεώρησης ε, σε όλους τους κρίκους της ε, αλυσίδα για να αποφύγουμε συσσόρευση του κέρδους σε ορισμένους μόνο κρίκους της αλυσίδα. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μέχρι τον Ιούλιο του 2018 έκθεση για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Πολλά λοιπόν μένουν να γίνουν, δεν είναι καθόλου εύκολο το πρόβλημα, είναι αρκετά δυσεπίλητο, αλλά τον Μάιο, συνεργασία με την Επιτροπή Προϋπολογισμών, εγκρίναμε κάποιες θέσεις και θα ξεκινήσουμε από τις 5 Ιουλίου τον τριμερή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι που θα μας δώσει ε, την ευκαιρία να αγγίψουμε τα θέματα, αλλά θα πρέπει να μας βοηθήσετε και εσείς στο Συμβούλιο, ώστε με τον κανονισμό Omnibus να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα πρόοδου και να αντιμετωπίσουμε ή να αναχαιτήσουμε αυτές τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Ευχαριστώ κύριο Ντές. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κυρία Υπουργό και τους κύριους Υπουργούς για την παρουσία τους εδώ. Και χαίρομαι που το θίγουμε το θέμα αυτό εκ γιατί το θέμα αυτό η Επιτροπή μα ε, το έχει συζητήσει επισταμμένο σε διάφορες περιστάσεις ε, και πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι καινούριο στο θέμα αυτό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες είμαι ε, πρόεδρος ε, επιτιμήσε μια ένωση συνεταιρισμού γαλακτοκομικού στην Βαβαρία και ξέρω τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο κόσμος. Και πέρσι, σε εποχές κρίσης, το κόμμα μας ε, και η πολιτική μας ομάδα έκανε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θα μπορούσε να την ε, λάβει υπόψη, να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να απαντήσουμε λοιπόν με νομοθετικές διατάξεις να αποτρέψουμε την υπερβολική συγκέντρωση η οποία ουσιαστικά δεν επιτρέπει την, ε, το ελεύθερο εμπόριο. Να σας υπενθυμίσω και τη συγκέντρωση υπάρχει στην Αυστρία και στη Γερμανία. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυτές οι μεγάλες τη παραγωγή έχουν και ίδια συστήματα πιστοποίηση. και θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πληρώνουν όλο και πιο πολλά οι mm-hmm. Δεν είναι όμως ε, καθήκον των ε, γαλακτοκομικών ε, επιχειρήσεων να ιδρύουν συστήματα πιστοποίηση. Είναι θέμα του κράτου και καθήκον του κράτου αυτό. τα θέματα επίση τη μονομερούς ε, καταγγελίας ε, των συμβάσεων. Το έχουμε ζήσει σε διάφορε περιστάσει αυτό. Να πέσουν τιμέ, δηλαδή και μονομερό να καταγγέλλονται οι συμβάσει. Ε, πρέπει αυτό νομοθετικά να ρυθμιστεί. Και επίση ένα θέμα που το έχουμε, το θέμα της, των τελών της μαφίας, όπως το αναφέρουμε στο κρατηδιό μου. Χρειαζόμαστε καθαρές, καθαρές τιμές γιατί υπάρχουν συστήματα εκπτώσεων όπου κανείς δεν έχει τελικά ε, αντίληψη και κανονική εντύπωση για το ποια είναι η τιμή. Θα πρέπει λοιπόν να είναι καθαρέ οι τιμέ για να υπάρχει διαφάνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό επίση. Ε, ο στόχο ε, σε ό,τι αφορά την προθεσμία πληρωμή χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ορίσουμε τι 30 ημέρε ω το όριο. Στην Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχει στον τομέα του κρέατο μια πρόθεσμια για την καταβολή των πληρωμών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει τέτοιο, τέτοια προθεσμία και κάτι άλλο που με εκνευρίζει ιδιαίτερω, ότι ο παραγωγό δεν εμφανίζεται στη συσκευασία. Έχουν οι μεγάλες ε, εταιρείε ε, τι δικέ του ε, υπηρεσίε συσκευασία και δεν εμφανίζεται πουθενά ο παραγωγό τελικά και είχαμε ζητήσει λοιπόν από την πλευρά τη πολιτική μου ομάδα να αναφέρεται ο παραγωγός. Τουλάχιστον σε εξίσου μεγάλα γράμματα, όπως και η εταιρεία. Και αυτό θεωρώ συμβάλλει στην γενικότερη διαφάνεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις σχετικές προδιαγραφές το 2004 και το 2005 Τότε που ξεκινήσαμε τη συζήτηση για τα τέλη περιαγωγής, πρέπει να σας πω ότι ήταν μεγάλη παρέμβαση στην ελεύθερη, στο ελεύθερο εμπόριο και πριν από λίγες ημέρες γιορτάσαμε επιτέλους την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Μα και εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να θυχτεί ξεκάθαρα, γιατί χωρίς η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα είχαν καταργηθεί και τα τέλη περιαγωγής. Και έτσι λοιπόν, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφέ προκειμένου να υπάρχει κάποιο περιορισμό για αυτέ τι μεγάλε αλυσίδε πλέον. Σα ευχαριστώ κύριε Νταντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω κυρία και κύριοι Υπουργοί για, για την παρουσία σας και για τις ομιλίες σας. Πριν από τέσσερα χρόνια ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη επισήμανε αυτή τη μάστιγα των αναθέμετων εμπορικών πρακτικών και την ασθενή θέση των γεωργών στην τροφική αλυσίδα και χαίρομαι για την πρωτοβουλία που αναλάβατε. Θα πρέπει να υπενθυμίζουμε να πάση στιγμή και προς τους πάντες ότι θα πρέπει να εξορροπήσουμε τα συμφέροντα των παραγωγών, των γεωργών και των καταναλωτών. Η κοινή γεωργική πολιτική έχει τουλάχιστον δύο Στόχου, όπως κατοχυρώνονται στις ε, συνθήκες. Θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπέ εισόδημα στο ίδιο παραγωγό και να προσπίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του καταναλωτή. Εμείς όμως στην Επιτροπή Γεωργία διαπιστώνουμε ότι η ερμηνεία που κάνουν οι αρχές του ανταγωνισμού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο έδωσαν περισσότερη έμφαση στα συμφέροντα ή τα ψεύδο συμφέροντα του καταναλωτή ε, και τα θεώρησαν υπέρτερα σε σχέση με τα συμφέροντα των καταναλωτών. Είχαμε 4 εκατομμύρια ανέργων το 2012 και εκεί ήταν 22% ε, η, η, ο προπολογισμό που αναφερόταν στα τρόφιμα. Τότε ε, αυτό ήταν πριν από πολλά χρόνια που δεν είχαμε τόσο τόση ανέργεια. Σήμερα όμως έχουμε πολύ περισσότερη ενέργεια 10%. Ε, και σίγουρα και ε, το τμήμα του προϋπολογισμού του νοικοκυριού που αφιερώνεται στα τρόφιμα είναι πολύ λιγότερο, θα πρέπει να αποκαταστήσουμε μια ισορροπία. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα πρώτα βήματα, όπως προβλέπει τον επίσημο έγγραφο, και είναι μια ε, μετριοπαθής αφετηρία, αλλά θα πρέπει να γίνει επιτέλους. Και μάλιστα στην Επιτροπή Γεωργίας ε, θα συζητηθεί αυτό το θέμα εντό λίγο. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε και εμεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια ξεκάθαρα μηνύματα για τη θέση μα. Γιατί προφανώ βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο και πραγματικά μπορούμε να ενισχύσουμε τη, τη θέση του παραγωγού. Αν πραγματικά ε, περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Γιατί φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή πλεύση. Ο κύριο Ερντό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχει περάσει πολύ ε, καιρό από τότε που τελείωσε η Σλοβακική Προεδρία και νομίζω ότι θα θέλαμε επευκαιρία να σας ευχαριστήσουμε για τις έξι μήνες εξαιρετικής εργασίας. Ε, θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί θα αλλάξω λίγο θέμα και θα θίξω ένα ζήτημα το οποίο ε, συνδέεται, αλλά όχι άμεσα ενδεχομένω. Χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τρεις υπουργούς ε, γεωργίας και έχω μια ερώτηση να σας θέσω και προς τους τρεις σας. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ επίκαιρο. η, ίδια συσκευασία, η ίδια επισήμανση, η ίδια διατροφική αξία μπορεί να υπάρχει, αλλά παρόλα αυτά ενδεχομένως να υπάρχει διαφορά στο περιεχόμενο ενός προϊόντος. Έγινε μια σχετική μελέτη στην Ουγγαρία και είδαμε μεγάλη διαφορά μεταξύ της ποιότητας των διαφορετικών προϊόντων. Πρόκειται λοιπόν για μια σοβαρή ανομαλία. Πώς μπορούμε να τη ρυθμίσουμε, με ποιο τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Σαντρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αναπόφευκτα θα επαναλάβω κάποια σχόλια που ήδη έγιναν. Ε, συμφωνώ και με τους υπουργούς, τους οποίους ευχαριστώ και θερμά για την πρωτοβουλία τους και για την παρουσία τους. Και πρόκειται για ένα θέμα που επισημαίνουμε εδώ και χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βρίσκεται στο επίκεντρο των οικονομικών θεμάτων και της αναζήτησης ισορροπίας και στη, γεωργία, και στη γεωργική οικονομία. Και συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες Ντεκάστρο, ε, Ντες και Νταντάν. Είναι Σημαντικό λοιπόν, ε, γιατί διαπιστώνουμε μία πραγματική συνένεση μεταξύ μας για τα θέματα αυτά και τον προβληματισμό μας. Θα πρέπει να βρούμε μία ισορροπία και στη θέση των γεωργών στην τροφική αλυσίδα. Εδώ και χρόνια το ζητούμε και το διεκδικούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η θέση του γεωργού στην τροφική αλυσίδα και χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να ανταποκριθούμε ε, στο θέμα αυτό και να λύσουμε το πρόβλημα. Επίση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλου του κρίκου τη αλυσίδα, τη τροφική αλυσίδα, γιατί μιλούμε εκτεταμένα για του παραγωγού και μα ενδιαφέρουν. Μιλούμε πολύ ιδιαίτερα για του διανομή, ε, τα σούπερ μάρκετ, αλλά μην ξεχάσουμε και τη μεταπητική βιομηχανία, που είναι ένα ενδιάμεσο κρίκο. Θα πρέπει να βρούμε ισορροπία μεταξύ όλων των κρίκων τη αλυσίδα. Χρειαζόμαστε μεν ευρωπαϊκά μέτρα, αλλά δεν αρκούν. Γιατί το θέμα του ελέγχου των αγορών σε διεθνέ επίπεδο επίση είναι κέριο και θα αποκτήσει πρωταρχική σημασία και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη τις λύσεις που θα προτείνουμε. Ναι, λοιπόν, ισορροπία, ναι, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος των γεωργικών αγορών και διεθνώς, παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Ντενανό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα της α, τροφικής αλυσίδας, το θε... η αλυσίδα σε τρόφιμα, είναι ένα περίπλοκο θέμα που επανέρχεται ξανά και ξανά. Και το Συμβούλιο Υπουργών και το Κοινοβούλιο καλό θα ήταν να προτείνει κάποιες πρωτοβουλίες και να ζητήσει την Κομισιόν να εγγύψει πιο σοβαρά στο θέμα. Ε, το θέμα του παραγωγού και το θέμα του καταναλωτή. Είναι σάκρε αλυσίδε, αλλά υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι κρίκοι. Και φυσικά και οι μεταποιητέ. Όταν βλέπω παραγωγού που γκρινιάζουν για τι τιμέ, ε, βλέπω και τους, ε, επίσης και τους μεταποιητές που γκρινιάζουν για τις, τιμέ, τιμές που τους επιβάλλουν μεγάλη διανομή, ε, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Είναι περίπλοκο το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να υπάρξουν περισσότερες ε, συμβάσεις. Οι παραγωγοί έχουν συμφέρον να ομαδοποιηθούν, να οργανωθούν σε συνεταιρισμού κτλ. Ε, και να δημιουργήσουν ε, ομάδε διαπραγμάτευση, όπω πρότεινε ο κ. Νταντά. Είναι σημαντικό να κινηθούν προ αυτήν την κατεύθυνση, ούτω ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν ειδικό βάρο απέναντι στου μεγάλου διανομή. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που το, που το θέμα της, του ανεφοδιασμού της, και των εστιατορίων Πώς θα, μπορέσουμε, πώς θα μπορέσουμε ούτως ώστε ε, τα σχολεία, ε, η και ε, να φτάνουν πιο γρήγορα κατευθείαν στον παραγωγό, ε, να αποφεύγουμε δηλαδή τις μεγάλες ε, αλυσίδες, να περνάμε από πολλούς μεταποιητές, ούτως ώστε ο καθένας να μπορέσει να καλύψει ανάγκες του. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό το θέμα. Και επίσης, για να ολοκληρώσουμε, νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα της σταθερότητα των τιμών. Το είπαν πάρα πολύ. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και το παράδειγμα που αναφέρατε κύριε Υπουργέ ε, για το τέλος της περιαγωγής είναι μια απόδειξη ότι όταν υπάρχει θέληση βρίσκουμε τη λύση όπως λέμε. Ε, καλό είναι να βρούμε τη θέληση ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια σταθεροποίηση των εισοδημάτων των γεωργών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σέχναλοβα. Ευχαριστώ τους υπουργούς. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρουσιάσετε τη θέση των χωρών σας. Εγώ είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η εσωτερική αγορά. Βασικά ε, δεν ήρθα εκτάκτος σε αυτή την Επιτροπή για να ακούσω την παρουσίαση αυτή του non-paper, ε, γιατί ασχολούμαι με την εσωτερική αγορά. Καλό θα είναι να υπάρξει και ένα έγγραφο της Επιτροπής Γεωργίας για τις αθέμητες γεωργικές πρακτικές και για τις εμπορικές σχέσεις. Ε, αυτό το non-paper περιγράφει πολύ σωστά αυτή την περίπλοκη σκέψη. Ε, όμως η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή ήταν η Επιτροπή ΙΝΚΟ στην πραγματικότητα όπου η συζήτηση έγινε πιο περίπλοκη και όλα αυτά καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το θέμα, να κάνουμε μια έκκληση προς το ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνει κάτι. Είμαι πεπισμένη ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο επιτροπές, την Επιτροπή Γεωργίας και την Επιτροπή ΙΜΚΟ, ήταν χρήσιμη για να εκπονηθεί τελικά αυτό το non-paper. Και θα ήθελα να γίνει και μία ακρόαση, αν γίνεται, και εδώ, αντίστοιχη με αυτή που κάναμε εμείς στην ΙΜΚΟ, ε, που ασχολήθηκε και με αυτό το θέμα και με την προστασία των καταναλωτών. Νομίζω ότι θα καταλάβουμε ακόμα καλύτερα την κατάσταση. Το ανεπίσημο αυτό έγγραφό σα περιγράφει πολύ καλά την κατάσταση. Μία, δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Προς την κυρία Ματέτσνα και προς τον κύριο Ντέιαν, που μιλήσαν για εθελοντικές πρωτοβουλίες είπαν και περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση. Θα ήθελα και ο κύριος Γιουρέσκα να μας πει δύο λόγια. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν αντίστοιχε δραστηριότητε και στη τεχική Δημοκρατία. Θα ήθελα να μα πει λοιπόν λίγα περισσότερα πράγματα. Με βάση τα όσα είπατε, 10 κράτη-μέλη στήριξαν το non-paper που ετοιμάσατε. Δηλαδή το ποτήρι αυτό είναι μισοάδιο μισογεμάτο, έτσι τελικά. Θα ήθελα να μου πείτε τι λείπει. ούτω ώστε να συμπαραταχθούν μαζί μας και άλλες χώρες. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έχετε τη στήριξή μας. Η έκπληξη έρχεται συνήθως από το Συμβούλιο. Επίσης, τα διπλά πρότυπα ποιότητα στο γεωργοδιατροφικό τομέα είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Καλό θα ήταν λοιπόν να γίνει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία πάνω στο θέμα αυτό. Επίσης, εγώ έκανα και μια νομική ανάλυση για το θέμα αυτό, ζήτησα να γίνει μάλλον, και καλό θα ήταν να υπάρξει και μια ειδική οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Νομίζω ότι θα μπορούσε να δοθεί συνέχεια λοιπόν σε αυτό το θέμα. Υπάρχει πάρα πολύ ψωμί εδώ. Κύριε Αγγιλέρα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις υπουργούς και να πω ότι οι απόψεις μας συμπίπτουν. Αυτή την αίσθηση έχουμε πάντως, της συνένεσης. Και εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας ε, έχουμε ξεκάθαρη θέση και φαίνεται και στο Συμβούλιο το ίδιο. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Επίτροπος Χόγκαν ε, έχει δεδηλωμένη και σαφή άποψη. Δεν ξέρω αν συμπίπτει με την άποψη της ε, ε, Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και του Επιτρόπου του Αρμόδιου για τον Ανταγωνισμό. Πάντως πιστεύω ότι έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε το μείζον πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, τις τιμές παραγωγού. Οι τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί για, το, για τη δραστηριότητά τους είναι απαράδεκτα χαμηλές. Και εγώ δεν πιστεύω στις εθελοντικές πρωτοβουλίες. Οι προαιρετικές πρωτοβουλίες και οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές, στην Ισπανία τουλάχιστον, δεν έχουν τελεσφορήσει. Δεν πιστεύω λοιπόν σε αυτή την οικειοθελή προσπάθεια, γιατί με τέτοιες εκούσιες πρωτοβουλίες τι κάνουμε ουσιαστικά, δίνουμε το πρόσχημα ε, στα κράτη-μέλη ή μια δικαιολογία που τη χρησιμοποιούν και τα σούπερ μάρκετ για να μην τις εφαρμόσουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που θα είναι η βάση της εναρμόνισης των εθνικών νομοθετικών διατάξεων. Χρειαζόμαστε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθετικό, ρυθμιστικό, ώστε οι 23, αν δεν κάνω λάθος, χώρες που έχουν θεσπίσει διατάξεις για τις θέμητες εμπορικές πρακτικές να τύχουν κάποιες εναρμόνισεις. Θα πρέπει να είμαστε πιο κατηγορηματικοί και αυστηροί για την αντιμετώπιση τους. Επίσης, είναι σημαντικό οι κυρώσει ε, να είναι ε, όχι συμβολικέ, αλλά πραγματικέ, για να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα και αποτέλεσμα. Πέραν όμω τη ε, ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι διατάξει που ισχύουν για τα όρια της συνεργασίας των ε, γεωργών. Να δούμε να διευκρινίσουμε τους, όμως τις διατάξεις μεταξύ τη κοινή γεωργική πολιτική και τη πολιτική ανταγωνισμού και θα πρέπει να υπερτερούν οι διατάξεις της ΚΑΠ έναντι των διατάξεων της πολιτικής ανταγωνισμού. Αυτό δεν είναι σαφές. Γιατί μερικές φορές είτε λόγω κοινοτική, εθνική ή περιφερειακή αρμοδιότητα, ε, λαμβάνονται απόψεις που έχουν, ε, θέσεις που των γεωργών. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τους κανόνες ανταγωνισμού και να ε, διευκρινίσουμε ότι υπερισχύουν οι διατάξει τη ΚΑΠ έναντι των διατάξεων του ανταγωνισμού. Είδε μη, θα τροφοδοτούμε ένα πυθμένο πηγάδι με, την, με τον προπολογισμό τη ΚΑΠ. Επίση, να τροποποιήσουμε τι διατάξει τη κοινή οργάνωση αγορά. Γιατί δεν εξυπηρετούν όλε οι διατάξει τη ΚΟΑ τον γεωργικό κλάδο. Θα πρέπει ή να τι διευκρινίσουμε αυτέ τι διατάξει τη κοινή οργάνωση αγορά ή να τις αναθεωρήσουμε. Αυτό περιμένουν οι Γεωργοί από μας. Εμπρός λοιπόν, να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συσπηρωθούμε, να ανασκουμποθούμε και να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση για να προστατεύσουμε τον κλάδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ροπέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπουργούς που ήρθαν εδώ σήμερα στη συνεδρίασή μας για να ακούσουμε και τις δικές μας απόψεις για το πώς το θέμα αυτό μπορεί να επιληφθεί. Φυσικά και χαιρόμαστε που υπάρχει καν αυτή η πρωτοβουλία και η Επιτροπή μας έχει συζητήσει τα θέματα αυτά σε διάφορες περιστάσεις στην τρέχουσα θητεία του Κοινοβουλίου. Έγινε και μια πρόταση για την επίλυση του ζητήματος. Και αλήθεια η απόφαση να είναι υποχρεωτική αυτή η λύση. Ωστόσο, μετά από τρία χρόνια το πρόβλημα δεν έχει ακόμα επιληθεί. Έχει οξυνθεί έτσι περαιτέρω. Και αυτό αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένα. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης και οι χώρες των παλαιών δημοκρατιών έχουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ παραγωγών και λιανεμπόρων. Τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέες δημοκρατίες αν θέλετε, βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση. Και είναι μάλλον ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Και όταν δεν υπάρχει λοιπόν η ιδιαίτερη πραγματευτική δύναμη από πλευρά των παραγωγών, οι μεταποιητέ και οι λιανέμποροι είναι αυτοί που τελικά υπαγορεύουν του όρου του παιχνιδιού. Όπως ανέφερε και ο υπουργό της Τσεχική Δημοκρατίας, 38% ξέρουμε ότι όταν έχουμε επιδοτήσεις πέφτουν οι τιμές. Αλλά αυτό δεν ε, είναι βιώσιμο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά το επιθυμεί, μπορεί να ρυθμίσει την κατάσταση. Για παράδειγμα, καταφέραμε να ρυθμίσουμε το τραπεζικό κλαμπ. Φυσικά και μπορούμε να βρούμε λύσει και στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά πολλά μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι οι συντονιστέ, τα κρατή-μέλη, μέσω διοργάνωση συνεταιρισμών και ενώσεων παραγωγών ή ενώσεων ανακλάδο. Αλλά προφανώ δεν μπορούν να τα κάνουν όλα τα κρατη από μόνα του και οι ίδιοι η παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει και κάποιε κανόνε και κάποιε γενικέ αρχέ για να εγγυάται κάποια δικαιώματα στα κρατη προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσει ανάλογα με τα ιδιαίτερα τη κάθε χώρα, γιατί είναι διαφορετική η κατάσταση στην Σουηδία από την Πορτογαλία, από τι βαλτικέ χώρε. Σα ευχαριστώ λοιπόν όλου και πιστεύω ότι από κοινού θα πετύχουμε αποτέλεσμα στο το τέλο του τρέχοντο έτου. Ο κύριο Μπούντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώ ήρθατε κύριε και κύριοι Υπουργοί. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και μας προβληματίζει όλους. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα καταπολεμήσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Αυτό είναι ιδιαίτερα φλέγο ζήτημα στις ε, χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε μια ομοιόμορφη ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θέμα αυτό. Δυστυχώς όμως ε, ε, διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη θετούν ε, διαφορετικέ λύσεις. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία πέρυσι εγκρίθηκε νομοθεσία που ρυθμίζει την προμήθεια γεωργικών προϊόντων την πώληση γεωργικών προϊόντων προς τους καταναλωτές. Και προβλέπει ότι τα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να διατίθενται σε προσιτές τιμές καταναλωτή. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία σε παραβάση κατά της Ρουμανίας λόγω αυτής της νομοθεσίας. Εξέτασα και προσωπικά αυτό το θέμα και πιστεύω ότι οι χώρες έχουν το δικαίωμα να προβλέπουμε τέτοιες βάσεις τη βραχυπρόθεσμη διάθεση γεωρικών προϊόντων. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Φυσικά και οι γεωργοί χρήζουν προστασίας και εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας στηρίζουμε τους γεωργούς αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα των καταναλωτών που θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν ε, τα εμπορεύματα που χρειάζονται σε προσιτές τιμές. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων αυτών. Ο κύριος Έρντος μας επισήμανε τα προβλήματα που υπάρχουν στις ανατολικές κυρίως χώρες με την ύπαρξη διπλών μέτρων και σταθμών για τα ίδια προϊόντα που έχουν διαφορετική ποιότητα ανάλογα με το που διατίθενται στη Δυτική Ευρώπη ή στην Ανατολική γιατί διαπιστώνουμε ότι ακόμη και στην ποιότητα των μηχανημάτων που πουλούνται στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν διαφορές, είναι ίσονος ποιότητα σε σχέση με τα ίδια μηχανέ τα ίδια μηχανήματα που πουλούνται στην Δυτική Ευρώπη. Ευχαριστώ, κυρία Μαγκίνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ του τρει υπουργού μα ε, που βρίσκονται εδώ σήμερα και πραγματικά πιστεύω ότι τέτοιου είδου ανταλλαγέ απόψεων χρειαζόμαστε πιο τακτικά, όχι μόνο με του υπουργού αλλά και με τα εθνικά κοινοβούλια. Σα ευχαριστώ λοιπόν που είσαστε εδώ σήμερα και σα ευχαριστώ και για την πολύ συνοπτική σα παρουσίαση. Να ευχαριστήσουμε και τη Σλοβακική Προεδρία για τη δουλειά που έκανε τον Ιούνιο του 2016. 600 μέλη του Κοινοβουλίου μα πλήρης ψήφισαν υπέρ της έκκλησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου. Είναι πολύ σαφής λοιπόν η τοποθέτησή μας και εσείς μας βοηθάτε να το πετύχουμε αυτό με το έγγραφο αυτό, το non-paper το οποίο μας παρουσιάσατε. Ξέρουμε ότι είναι πολύ περίπλοκος ο τομέας, ο κλάδος αυτός και αν θα μπορούσαμε να δώσουμε λίγο να κατανοήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την κατανοούμε γιατί είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να απαιτήσουμε να η δράση. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο θέμα τη περιαγωγή, των τέλων περιαγωγή. Ελπίζω να μην χρειαστεί και τόσο πολύ χρόνο για να περάσουμε αποτελεσματική νομοθεσία στον τομέα αυτό, όπως στον τομέα τη περιαγωγή. Ωστόσο, σε κάποιε περιπτώσει χρειάζεται και πίεση και χρειάζεται και χρόνο για να πετύχουμε ένα στόχο. Αλλά θεωρώ ότι το πλαίσιο είναι ευρύτερο από αυτό που παρουσιάστηκε στη συζήτηση. Το θέμα τη χρηματοδότηση και του προπολογισμού είναι σημαντικό. Αλλά πέραν τούτου έγινε και μια συζήτηση για την αλλαγή του κλίματο την προηγούμενη εβδομάδα και τι σημαίνει αυτό στην γεωργία και πώς θα πρέπει να αντιδράσει ο κλάδος αυτός. Έγιναν πολλές συζητήσεις για τα δημόσια αγαθά και το ότι η γεωργία θα πρέπει να κάνουν πιο πολλά για το περιβάλλον και την βιοπικιλία. Αν συνεχίσουμε λοιπόν, αν συνεχίσει η πίεση στην τετραφική αλυσίδα, στην αλυσίδα διατροφική παραγωγής, όπως υπάρχει σήμερα, πολύ φοβάμαι ότι θα αποτύχουμε σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, γιατί οι γεωργοί θα πρέπει να μπορούν να επενδύουν και μπορεί κανείς να επενδύσει. Μπορεί να του περισσεύει και κάτι για να το επενδύσει, πρέπει να ζει και να του περισσεύει και κάτι για να το επενδύσει. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις όμως οι αγρότες ε, επιβιώνουν, δεν επενδύουν δε. Και θα πρέπει λοιπόν κάπως να αντισταθμίσουμε αυτή την έλλειψη επενδύσεων, την έλλειψη αν θέλετε κέρδους. Έχετε την υποστήριξή μου για το θέμα αυτό και να σας πω την αλήθεια έχουμε ήδη ξεκινήσει το 2005 τη συζήτηση αυτή, σχεδόν όσο και για τα τέλη περιαγωγή έχει πάρει στη συζήτηση. Αλλά καλό θα ήταν, πιστεύω, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξουμε τι βέλτιστε πρακτικέ σε επίπεδο κρατών μελών. Να μην χρειαστεί να επανεφεύρουμε τον τροχό ενωμένοι πιστεύω μπορούμε να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαλύνει αν θέλετε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των επιτρόπων στο θέμα αυτό γιατί υπάρχουν διαφορές και να ακολουθήσει τον δρόμο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαρνιού. Είπε η κυρία Μαγκίνης ότι 600 ευρωβουλευτές ε, ψήφισαν ε, υπέρ. Εγώ δεν ήμουν ένα από τους 600. Να, θέλω το ξέρετε όλοι σα. έτσι. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε αυτό το πρόβλημα. Εδώ και καιρό. Ε, με τους στενοπολιτές. Και η λύση μας ήταν να διοργήσουμε ένα διαμεσολαβητή για τα σούπερ μάρκετ. Η Κρίστιν ε, είναι η διαμεσολαβήτρια από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η θέση και η οποία σιγά σιγά αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Το 2015 στηλίτευσε ε, στυλίτευσε την Τέσκο που είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί καθυστερήσε τις πληρωμές στους προμηθευτές. Αυτή η κατηγορία ας πούμε ε, ήταν πάρα πολύ καλή διότι ήταν πολύ καλή τεχνική διότι δεν τους αρέσει η κακή δημοσιότητα. Επίσης, ε, την ίδια χρονιά της δώσαμε τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις ε, στους, στα σούπερ μάρκετ που ήταν το 1% του κύκλου εργασιών. Αλλά όμως ασχολείται μόνο με τους λιανοπολιτές, ε, σούπερ μάρκετ κτλ. και τους προμηθευτές τους. Εάν υπάρξει αυτό το σχήμα, βλέπω τα εξής προβλήματα. Ε, υπάρχει, ε, αν υπάρχει δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι αντίστοιχο, μπορείτε να μα δημιουργήσετε προβλήματα σε εθνικό επίπεδο. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτά που λειτουργούν σε εμά. Και επίση, ακούσαμε ομιλητέ να λένε σήμερα ότι υπάρχουν διαφορετικέ συμπεριφορέ ε, στο εμπόριο σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε. Και ένα φίλο μου, ο οποίο ε, δίνει μηχανήματα στη Γερμανία και στην Ιταλία, λέει ότι αυτέ οι δύο χώρε λειτουργούν τελείω διαφορετικά. Και η Ρουμανία, α πούμε, είναι ακόμα χειρότερη περίπτωση ε, είναι πολύ πιο διαφορετική. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε ένα ευρωπαϊκό σχήμα παντού, σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω θα υπάρξει μεγάλη ε, αντίσταση και μνησικακία. Ε, επίσης, όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να συλλέγονται κεντρικά. Ε, ξέρετε βέβαια πόσο καλή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρτούρα. Ε, μπορεί να χρειαστούν χρόνια πριν να εφαρμοστεί αυτό το έγγραφο. Και τέλος, επίσης, ε, θα υπάρξει διαφθορά, προφανώς. Ε, όταν έχουμε αυτούς τους μεγάλους παίχτες στα σούπερ μάρκετ, μπορεί κάλλιστα να διαφύρουν με δωροδοκία τους επιτρόπους, έτσι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε διάφορες γεωργικές επιχειρήσεις, μεγάλες, μεγάλους παραγωγούς, ε, μεγάλους παραγωγούς, ας πούμε, πατάτας, καρότων, πουλερικών, αυγών, κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Όσοι παράγουν αυτά τα προϊόντα έγιναν όλο και ή έγιναν μεγαλύτεροι, μεγενθήθηκαν ή βγήκαν από την αγορά. Οι μεγάλοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις συχνά αυτών που έφυγαν από την αγορά. Συχνά, ας πούμε, ε, ε, πατάτες να καλλιεργούνται σε μια α, γεωργική εκμετάλλευση που δεν ανήκει α, σε αυτόν που καλλιέργεια τη πατάτε, α πούμε. Αυτό που έχει τη γη, α πούμε, νοικιάζει τη γη του και χρησιμοποιεί ο άλλο τα μηχανήματα κτλ. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το ρολόι πίσω, έτσι. Ε, για να δούμε λοιπόν πού θα μα οδηγήσει το μέλλον. Ο Σε Εδώ, ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα από πλευρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ του ε, υπουργού και ιδιαίτερα τον ε, Σλοβαίνο υπουργό, τον υπουργό μα ο οποίος εδώ και κάποια χρόνια είναι γνωστός στην Σλοβενία και εδώ α, άλλωστε για τον αγώνα που δίνει για το θέμα αυτό και έχει πετύχει και κάποια αποτελέσματα στον κλάδο αυτό. Τα αποτελέσματα αυτά όμως δεν είναι ακόμα εμφανή, όχι αρκετά. Ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή μας σήμερα. Είμαστε σύμμαχοί σας, μιλούμε την ίδια γλώσσα. Και εδώ είναι το σωστό σημείο για να ανταλλάξουμε πρακτικές και να πετύχουμε κάτι. Και ακόμα και είναι δύσκολο να πείσουμε του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν κάτι για τον κλάδο αυτό. Τέλη του έτου είχαμε την παρουσίαση τη έκθεση την οποία είχε αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Επιτρόπου Χόγκαν και αυτή η έκθεση είπε ξεκάθαρα κατάφερε, μάλλον κατέληξε στο εξή πόρισμα, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση έτσι. Μπορεί ορισμένοι να μην θέλουν να υπάρξει παρέμβαση στην νομοθεσία, αλλά ιδάλω δεν θα ρυθμιστεί η κατάσταση. Και χαίρομαι που μεταξύ των προσυπογραφούντων είναι και επτά υπουργοί από κράτη της ε, Βαλτικής. Ε. Περιλαμβάνεται λοιπόν μια σαφή ανάλυση της κατάστασης και των τάσεων που διακρίνονται και είδαμε ότι στα κράτη ακριβώς αυτά η κατάσταση είναι πιο δύσκολη από ότι στα παλιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει πιο ελλειπής οργάνωση της ε, Γεωργίας. Ξέρουμε ότι ασφαλώς υπάρχουν ε, ιστορικά προβλήματα με τους συνεταιρισμούς. Και όταν μελετήσαμε την οργάνωση της οικονομίας, διαπιστώσαμε είδαμε ότι ένα μεγάλο τμήμα της του κλάδου δεν είναι καν οργανωμένο. Και ότι η οργάνωση αυτή έγινε σε μετάπιτα χρονικό σημείο. Το πρόβλημα ενδεχομένω να επιληθεί από την πιο ισχυρή υποστήριξη των αγροτικών ενώσεων. Και στην μπραντική λοιπόν γεωργική πολιτική θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στα θέματα αυτά και ενδεχομένω να λάβουμε και κάποια μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. στη συνέχεια. Υπάρχουν αυτές οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ε, η συγκέντρωση για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις γεωργικές αγορές. Είδαμε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι τόσο ασχήμη στην κατάσταση αυτή που πραγματικά θα πρέπει να παρέμβουμε. Αν ήταν δυνατόν να παρέμβουμε στην ενεργειακό κλάδο, όπου οι εταιρείε υποχρεούνται να πληρώσουν πρόστιμα, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε και κάτι αντίστοιχο στον κλάδο αυτό. Οι καταναλωτές λοιπόν θα είναι αυτοί που θα νιώσουν και τη διαφορά επίσης και θα πρέπει να υπάρχει θέληση οργάνωσης. Αν οι καταναλωτέ, επαναλαμβάνω, ασκήσουν πίεση για την διοργάνωση στο επίπεδο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις υπουργούς που ήρθαν εδώ σήμερα. Δεν μας συμβαίνει τόσο συχνά να βλέπουμε τέτοια υψηλή εκπροσώπηση. Αλλά του ευχαριστώ επίσης και για την ευαισθησία που δείχνουν απέναντι σε αυτό το θέμα, που είναι πολύ σημαντικό θέμα για το γεωργικό κλάδο. Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημασία της σωστής λειτουργίας του κλάδου, του διατροφικού κλάδου, της διατροφικής αλυσίδας και επίσης είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι η γεωργή είναι ο αδύναμος ε, κρίκος αλυσίδας. Η ΚΑΠ ε, δίνει εργαλεία για να ενισχύσουμε τη θέση των ε, Ευρωπαίων γεωργών, αλλά αυτά τα εργαλεία φυσικά δεν χρησιμοποιούνται το ίδιο αποτελεσματικά σε όλες τις χώρες και σίγουρα πρέπει να βελτιωθούν. Πρέπει να βρεθούν λύσεις για να εγγυηθούμε ότι οι κίνδυνοι μοιράζονται πολύ πιο δίκαια σε όλη την γεωργοδιατροφική αλυσίδα και ότι το κίνητρο των συμβάσεων βελτιώνεται, βελτιώνεται η διαχείριση της αγοράς και η διαχείριση των κινδύνων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυστυχώς νομοθετική πράξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να αντιμετωπίσει τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές των διαφόρων φορέων της τροφικής αλυσίδας. Ένα πρώτο βήμα έγινε με το Omnibus και ευχαριστούμε τον, ε, τον κύριο Ντέσε και τον κύριο Ντεκάστρο, του συζητητέ που είχαν αυτή την ευαισθησία για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί, πρέπει να κάνουμε και κάτι ακόμα. Και εμεί είχαμε παρουσιάσει μία πρόταση για μία πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία δέχτηκαν νομίζω όλοι, συνολικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί του θέματος αυτού. Η πρόταση είναι να ζητήσουμε από την Κομισιό να υποβάλει πρόταση ούτως ώστε να βελτιωθεί η ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τον τρόπο αντιμετώπισης των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Η Οδηγία 29 του 2005 δηλαδή, ούτως ώστε να ενταχθεί και το πρόβλημα των αθέμητων γεωργικών πρακτικών στο πώς αντιμετωπίζουμε τον, την τροφική αλυσίδα. Επίσης, ε, οι όροι ανταγωνισμού θα πρέπει να δημιουργήσουν προθέσεις ε, για μια πιο δίκαιη αγορά, ούτως ώστε ο καταναλωτής να υποφελείται από μια ευρύτατη αλυσίδα ε, καλών προϊόντων με ανταγωνιστικές τιμές και επίσης να δίνονται κίνητρα για επενδύσεις χωρίς να περιορίζονται οι παράγοντες της αγοράς λόγω αυτών των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Υπάρχει μια γενικευμένη ευαισθησία, όλοι συζητήσαμε που, που είμαστε εδώ σήμερα, μιλάμε όλοι υπέρ της προστασίας των συμφερόντων. Τώρα, καλό είναι από τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη, περιμένουμε γρήγορα μια πρόταση για μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ο κύριος Νέκοφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τους τρεις υπουργούς που ήρθαν στην Επιτροπή μας και μας παρουσίασαν την πρωτοβουλία τους. Οι συνάδελφοι επέμειναν ε, στην ανάγκη εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και ίδιας ποιότητας ε, ανεξάρτητα από το που πολλούνται τα προϊόντα. Και σίγουρα χωρίς ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο τίποτα δεν θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε. Ερωτώ λοιπόν ε, τους εκπροσώπους των ε, αλυσίδων διανομής. Ε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αδυναμίες στην ε, τροφική αλυσίδα, σε διάφορους κρίκους αλυσίδας. Αλλά φαντάζομαι οι αλυσίδες διανομής θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένες γιατί είναι οι προνομιούχες της τροφικής αλυσίδας. Παρόλα αυτά, στην Βουλγαρία υπάρχει πρόβλημα και στον κλάδο της διανομής. Και πολλοί διανομής παραπονιούνται. Μιλούμε για αύξηση της, ε, του παγκόσμιου πληθυσμού και την ανάγκη να συστήσουμε ολόκληρη την ανθρωπότητα και άρα ανάγκη αύξηση της γεωργικής παραγωγής και των γεωργικών προϊόντων. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη θέση των γεωργών. Πώς είναι δυνατόν ε, να επιβιώσουν οι γεωργοί μας όταν... Ε, τα εισοδήματά τους δεν, δεν τους εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Πώς θέλουμε λοιπόν να στήσουμε την ανθρωπότητα όταν ε, τα μέτρα μας βοηθούν τις αλυσίδες διανομής ε, και όχι τους γεωργούς και άρα τους δίνουν ενάβσματα να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και να ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τους συναδέλφους που σας καλωσόρισαν εδώ στη σημερινή συνεδρίαση, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή το ότι έχουμε μαζί μας τρεις υπουργούς από λίγο πολύ την ίδια περιοχή, από νέα κρατημέλη και οι τρεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με αυτά που ακούσαμε από τους συναδέλφους. Διάβασα πάρα πολλά άρθρα πραγματικά και έκανα και πολλές διαβουλεύσεις αλλά με πάσα ειλικρίνεια δεν είδα καμία επιστημονική βάση ή ανεξάρτητη έρευνα επί του θέματος αυτού. Καταλαβαίνω ότι τα διάφορα όργανα και διάφορες υπηρεσίες ε, ανακυκλώνουν λίγο πολύ, ενδεχομένως εθελημένα, αυτά που τους συμφέρουν και θέλουν να ακούσουν, αλλά αναρωτιέμαι κατά πόσον έχετε οποιοδήποτε επιστημονικό υπόβαθρο σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατών μελών. Ένα δεύτερο θέμα. Πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα. Και ο ΦΠΑ αποτελεί συνήθω και συχνά ένα εργαλείο για θέμη την εμπορική πρακτική. Υπάρχει μεγάλη κερδοσκοπία, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ ακόμα και κίνδυνος θα έλεγα σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ. έξω. σου κατάλαβα όμως, ε, μερικοί εξημών έχουν ε, εμπειρία σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ στα γεωργικά προϊόντα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την ε, άποψή σας για το θέμα αυτό. Τρίτο ζήτημα, και εδώ θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο τον κύριο Μπόκοβιτς, με τον οποίο προσπαθούμε να πρωτοστατήσουμε για κάποια έργα σε ό,τι αφορά και ε, το πρόγραμμα των αφιών ε, περιφερειών. Δεν θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να βοηθηθούν οι μικρές ε, κοινότητες της υπέτρου προκειμένου να συμμετέχουν στον σύγχρονο κόσμο. Και επίσης, τι πιστεύετε για το μέλλον της ε, Γεωργίας. Ο κύριος, η κυρία Πτήρη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους υπουργούς που ήρθαν στη συνεδρίασή μας. Ε, με βάση την ε, Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός από τη Δανία και τη Σουηδία, οι υπόλοιπε χώρες μέλη έχουν ε, εθνικές νομοθετικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Μερικές ε, είναι γενικού χαρακτήρα και άλλες πιο ειδικού χαρακτήρα. Ε, φυσικά θα πρέπει να φροντίσουμε τους Γιώργους μας, να μην χρειάζεται να φτάσουν να ζητιανεύουν ή να φτάσουν στο χείλο της χειροκοπίας και γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε μέτρα και όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και στηρίζω ολόθερμα την πρωτοβουλία σας για ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αντιμετώπιση αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Εγώ κατάγομαι από την Κροατία και μπορώ να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένη που θέτεται αυτό το θέμα σημαντική πρωτοβουλία και μάλιστα έγινε δεκτή και η δική μου πρωτοβουλία να ε, θεσπιστούν και στην Κροατία νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αθέμητων εμπορικών πρακτικών, γιατί η προηγούμενη προσέγγιση δεν απέφερε καρπούς. Επίσης, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω για μια πρακτική που διαπιστώνουμε για την ε, διαφορά στην ποιότητα δηλαδή των ίδιων προϊόντων ανάλογα με το αν πολλούνται στη Δυτική στην Ανατολική Ευρώπη. Και μάλιστα υπάρχουν έρευνες ε, που τεκμηρώνουν αυτή τη διαπίστωση έγιναν συγκρίσεις ε, για τα ίδια προϊόντα μεταξύ Σλοβενίας και Αυστρίας και των προϊόντων που διατίθεται στη Γερμανία και στην Κροατία. Οι έρευνες ε, διαπίστωσαν διαφορά στην ποιότητα για τα ίδια προϊόντα ανάλογα με το που πολλούνται. Είναι σημαντικές ε, λοιπόν οι απάτες αυτές ουσιαστικά που βάλουν κατά των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθούν ευρωπαϊκά μέτρα και αυστηρές κυρώσεις για τέτοιου είδους απάτες. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι αρνητικό και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι θετικό για να προσελκύσουμε και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προτάσεις της να θέσει ένα τέρμα σε τέτοιες διακρίσεις βάρος των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σας ευχαριστώ κύριο ε, thank you very much. Ε. Ευχαριστώ. Χάρη στο θαύμα της τεχνολογίας, ε, άκουσα, άκουγα αυτή τη συζήτηση, ενώ ήμουν αμπλεγμένος σε κυκλοφοριακή συμφόρηση. όταν είναι κάνει σε κυκλοφοριακή συμφόρηση και όλα κινούνται πάρα πολύ αργά, βλέπω ότι αλλού όλα κινούνται με αγαστή συνεργασία. Κοιτάξτε, ε, τα τελευταία τρία χρόνια ε, πριν από τις τελευταίες εκλογές ε, συζητάμε συνέχεια αυτό το θέμα, προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις κτλ. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει το πρόβλημα των αθέμπτων εμπορικών πρακτικών, είμαστε σίγουροι ε, και έχουμε παραδείγματα και τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί τελικά, εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, το πιο σημαντικό, ο πιο σημαντικός κρίκος στη διατροφική αλυσίδα που είναι οι γεωργοί θα χάσουν εάν δεν τους βοηθήσουμε. Ε, και επίσης θα υπάρξει και, και καμία ανανέωση. Κανένας δεν θα θέλει να γίνει γεωργός πια. Εάν δεν έχεις καλές τιμές για την προσπάθειά σου, δεν παίρνεις καλές τιμές, γιατί να γίνεις γεωργός. Ε, όσο έχουμε το Δαβίδ και το Γολιάθ, ε, κοιτάξτε, ε, και ενώ στη βίβλο, ας πούμε, ο μικρός σκοτώνει ο Δαβί σκοτώνει τον Γολιάθ. Ε, εδώ πέρα δεν συμβαίνουν στην πραγματική ζωή αυτά κάθε μέρα, αυτά τα θαύματα. Έτσι. Οι μεγάλοι πρέπει κάπω να περιοριστούν, έτσι, ούτω ώστε η μάχη να είναι λίγο πιο ισότιμη. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ε, ίσως σε πανευρωπαϊκή ε, νομοθεσία. Εάν όλοι συνεργαστούμε μαζί, ε, γιατί ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται ε, συχνά προσπαθούν να βρουν παραθυράκια μέσω των διεξόδων που τους δίνει η εθνική νομοθεσία. Αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια αν το συζητάμε θεωρητικά. Έτσι. Και όσο θεωρητικολογούμε τόσο πιο πολύ καθυστερούμε τη δράση. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ας ανασκουμποθούμε επιτέλους. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ο Διευθυντής ΧΑΠΣ. Ευχαριστώ. Σας Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως την ε, Υπουργό κυρία Τιματέτσνα για την δουλειά που έκανε και αυτή και η ομάδα της πέρσι κατά το δεύτερο ήμιση του 2016. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερη η επιτυχία το ότι καταφέρατε να συμφωνήσουν 28 κράτη-μέλη για τα πορίσματα του Συμβουλίου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό ως ε, αποτέλεσμα και το πετύχατε. Το συζητήσαμε και σήμερα το απόγευμα. Το πρόβλημα είναι ότι οι αθεμίδες εμπορικές πρακτικές αποτελούν ένα πάρα πολύ περίπλοκο και ευρύτερο θέμα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν ούτε οι ίδιοι όροι, ούτε οι ίδιες βάσεις στα κράτη-μέλη και αυτό προκαλεί μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες. Πολλά κράτη-μέλη πολύ απλά δεν έχουν και τη διάθεση να νομοθετήσουν η οποία θα χρειαζόταν στη τελική ανάλυση, πιστεύω ότι το non-paper το οποίο παρουσιάσατε αποτελεί και ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, και απόρρια των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε στο Συμβούλιο για την επιτευξή συμφωνίας, γιατί το νόμο paper πάει και παραπάνω και παραπέρα από τα πορίσματα του Συμβουλίου. Από την άλλη υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο μετράει ιδιαίτερως ε, για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το ψήφισμα με τις 600 ψήφου, ψήφους υπέρ της προώθησης των νομοθετικών προτάσεων. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα μας βοηθήσει να προωθηθεί αυτή η διαδικασία. Όλοι γνωρίζουμε ότι το γεγονό ότι υπάρχουν αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ αφέ αυτού αποτελεί ένα δείγμα του ότι η αγορά δεν λειτουργεί όπω θα έπρεπε. Δεν λειτουργεί σωστά και όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία και να φροντίσουμε το τι γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Να κινηθούμε με μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο. Υπάρχει δε και η μεγάλη ευκαιρία αύριο που θα παραβρεθούν ε, εδώ οι δύο αρμόδιοι επίτροποι και είμαι βέβαιος ότι ο Επιτροπός Βέστριγκαρτ και ο Επιτροπός Χόγκαν θα παρουσιάσουν κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να προωθήσουν την διαδικασία προς τη σωστή κατεύθυνση επί του παρόντος. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. και προσβλέπω και στην αυριανή συζήτηση εδώ στην Επιτροπή σας. Σίγουρα θα είναι ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο και πάλι στους καλεσμένους μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε καλεσμένους ε, από ε, κοινοβούλια διαφόρων χωρών του κόσμου μετά από πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης ΕΞΠΟ, Εξωτερικών Πολιτικών, στα πλαίσια του προγράμματος ε, ε, ε, στήριξης της δημοκρατίας. Σας καλωσορίζουμε θερμά τους βουλευτές από διάφορες χώρες του κόσμου. θα διαπιστώνετε ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για πολλές χώρες, το θέμα που συζητούμε σήμερα. Θα δώσω τώρα και πάλι το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν θα πρότεινα με την ίδια σειρά που τους ακούσαμε και προηγουμένως. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ και για τη στήριξη που εκφράσατε. Είναι σαφές ότι εμείς όταν υιοθετήσαμε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας τα συμπεράσματα με ομοφωνία, Είχαμε τονίσει εμεί από πλευρά Προεδρία ότι δεν σκοπεύουμε καθόλου μετά την υιοθέτηση των συμπερασμάτων να εγκαταλείψουμε τη μάχη. Είναι άνθρωποι οι Γεωργοί που θέλουμε να προστατεύσουμε. Είναι προτεραιότητά μα. Είναι σημαντικό το γεγονό ότι αποφασίσαμε για αυτά τα πράγματα ω εμεί οι Υπουργοί Γεωργία και Ανάπτυξη Πέθρου. Νομίζω ότι η γεωργία γενικά είναι ένα κλάδο που πρέπει να προστατευτεί. Πραγματικά ένα συνάδελφο είπε ότι είναι μία μάχη ανάμεσα στο Δαβί και στο Γολιάθ. Έτσι είναι, πραγματικά. Ε, οι μεγάλοι διανομή, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν στα χέρια του ένα τεράστιο κεφάλαιο και είναι δύσκολο να του ανταγωνιστεί κανεί. Παρότι νομίζω ότι ο κύριος Ντες μίλησε για κάποιες οργανώσεις παραγωγών που κάνουν καλή δουλειά, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανείς τις γνώσεις, τις οικονομικές, νομικές κτλ. για να αντιμετωπίσει αυτού τους μεγάλους διανομή. Είναι σημαντικό λοιπόν για να κάνουμε κάτι, να έχουμε μια νομοθεσία για να ρυθμίσουμε τον τομέα. Έχουμε ρυθμίσει τις τηλεπικοινωνίε, την ενέργεια, το νερό, γιατί όχι τη γεωργία. Το αξίζει. Σα ευχαριστώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη, για τον ενθουσιασμό και ελπίζω στο εγγύς μέλλον να καταφέρουμε να προχωρήσουμε αυτή την πρωτοβουλία και να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Εκτιμώ πάρα πολύ τις ε, παρεμβάσεις σας, όλους εσάς που μας στηρίζετε στην προσπάθεια που κάνουμε. Ακούσαμε διάφορα, διάφορες παρεμβάσεις, επιχειρήματα, από Βρετανούς ε, ευρωβουλευτέ, αλλά και από άλλου που εξέφρασαν κάποιε ανησυχίες. Να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ακούσει ποτέ να γίνεται λόγος για εθελοντική περιαγωγή. Κάποια στιγμή καλό, ήταν, καλό θα ήταν, ή μάλλον, φανταστείτε, ότι η Κομισιόν κάποια στιγμή λέει «Α, κοιτάξτε, κάντε μια θελοντική προσπάθεια, ε, δώστε μας αυτό το, αυτό το roaming σε χαμηλές τιμές, ας πούμε, χρησιμοποιήστε τον, τα δίκτυα που υπάρχουν, αλλά ε, κατεβάστε την περιαγωγή». Υπάρχει τέτοια περίπτωση ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή η εθελοντική προσπάθεια. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τιμές ε, που δίνουμε στους παραγωγούς, ε, που δεν καλύπτει καν το κόστο τους. Ε, πρέπει να βοηθήσουμε τους γεωργούς. Δεν έχει νόημα να πιστεύουμε, είναι αφελές να πιστεύουμε ότι θα κάνουν κάτι από μόνοι τους οι μεγάλοι διανομής. Προς το Βρετανό συνάδελφο. Εγώ πήγα στη Βρετανία, όχι υπό την επίσημη ιδιότητά μου, και μίλησα με γεωργούς Βρετανούς. Υπάρχουν ε, φόβοι από πλευρά του ότι αν δεν ε, υπερασπιστούμε το Δαβίδ, θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια σε μια κατάσταση όπου οι μικροί γεωργοί, οι πικρέ ε, εκμεταλλεύσει θα εκμεταλλευτούν. Γιατί ο τοπικό παραγωγό, αν θέλει να διαπραγματευτεί με ένα μεγάλο διανομέα, τι του λένε. Πολύ ωραία, αλλά σου δίνουμε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή, ο όγκο των προϊόντων θα πρέπει να είναι σε ένα τάδε επίπεδο. Ε, θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να καλύψει ανάγκε τουλάχιστον τριών ή τεσσάρων ε, εκατομμυρίων κατοίκων. Ποιο μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, ποιο μπορεί να σεβαστεί αυτέ τι προποθέσει. Αν θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε την ύπεθρο και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει στο γεωργικό τομέα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώ. Αυτά και κλείνω. Και στρέφουμε, α, πριν κλείσω, ε, προς την Επιτροπή. Στα πλαίσια του non-paper, εμείς ε, περιγράψαμε όλες τις αθέμητες πρακτικές. Τις περιγράψαμε, φτάσαμε και σε συμπεράσματα, προτείναμε και λύσεις. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα η Κομισιόν σε λίγους μήνες να ετοιμάσει ένα νομοθετικό κείμενο απλό, ούτω ώστε να σταματήσουν πια αυτές οι αθέμητες ε, εμπορικέ πρακτικές. Ε, έρχομαι εδώ με ταπεινοφροσύνη, σας κάνω αυτή την πρόταση. Ελπίζω να μπορέσετε κάτι να κάνετε, γιατί Σίγουρα ε, καλό θα ήταν ε, να γίνει κάτι και θα σας ήταν ευγνώμονες η Γεωργία αν κάνετε κάτι. Σας ευχαριστώ κύριε Ζήταν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Θα επιστρέψω στην πατρίδα μου τη Σλοβενία πολύ πιο αισιόδοξο από ό,τι ήρθα. Γιατί διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο και αυτό μα δίνει περισσότερη φόρα και ενθουσιασμό να προχωρήσουμε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που επισημάναμε. Και διαπιστώσαμε ε, χειρότερη ποιότητα στα προϊόντα της Ανατολικής Ευρώπης σε σχέση με αυτά της Δυτικής Ευρώπης. Στη Σλοβενία δεν διαπιστώσαμε τέτοια διαφορά. Είναι αδύνατον να έχουμε τα ίδια προϊόντα σε δύο διαφορετικές χώρες και να είναι ίδιες ποιότητας. δεν είναι φυσιολογικό ε, ένα, το ίδιο προϊόν στη Γαλλία να είναι ανώτερη ποιότητα από το αντίστοιχο στη Σλοβενία ή στη Σλοβακία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε παρόμοια ποιότητα των προϊόντων όπου και αν διατίθενται. Επίσης, μιλήσαμε για αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Εγώ θα προτιμούσα να τις λέμε αθέμητες πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων γιατί υπάρχουν κάποιες αδικίες μεταξύ παραγωγών και διανομέων, αλλά δεν είναι οι μόνες αδικίες στην κρίση του γαλακτοκομικού τομέα. δεν χρεοκόπησε κανένας γαλακτοπαραγωγός, όλοι εξασφάλισαν τα περιθώρια κέρδους τους. Η γεωργοί ήταν αυτή που βρέθηκαν στη χειρότερη θέση και μερικοί κτηνοτρόφοι χρειάστηκε, η γαλακτοπαραγωγή χρειάστηκε να κλείσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Δεν επλήγησαν από τη γαλακτοκομική κρίση ούτε οι μεταπίτε ούτε οι διανομή. Επίσης μιλήσαμε για εθελοντικούς ε, κώδικες συμπεριφοράς. Δεν νομίζω ότι με εκούσιες πρωτοβουλίες θα επιτύχουμε τίποτα. Μπορούμε να το λέμε, αλλά αν επαφιόμαστε στην καλή θέληση του Α και του Β δεν πρόκειται να έχουμε εμφανή αποτελέσματα. Εξού και η πρότασή μας. Προτείνουμε νομοθετικές διατάξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έστω και αν αυτές περιορίζονται στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, σε ένα κοινό βασικό σημείο αφετηρία. Θα πρέπει να υπάρχουν παρόλα αυτά κάποια κοινά μέτρα και 27 χώρες να τηρούν τη μέγιστη περίοδο πληρωμής των 30 ημερών. Δεν θα πρέπει να καθυστερούν οι πληρωμές πάνω από 30 ημέρες και θα πρέπει να ισχύει αυτή η διάταξη ομοιόμορφα παντού. Επίσης θα πρέπει να επιβάλλονται ποινές πρόστιμα 1% του τζίρου, του κύκλου εργασιών. Τότε θα δούμε αν οι ευρωπαϊκές δράσεις λειτουργούν ή όχι. Ευχαριστώ κύριο Δέσης, ζήτησε και πάλι το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο, γιατί θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Ασχέτως Πολιτική ιδεολογία και σε ποια πολιτική παράταξη και ο καθένα στηρίξαμε αυτή την πρωτοβουλία των τριών υπουργών. Περιμένουμε τώρα μια νομοθετική πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί το 2004 ξεκινήσαμε την πρόταση για την κατάργηση των τελών περιαγωγή και χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να εφαρμοστεί και εμπράκτο αυτή η πρόταση. Και διαπιστώσαμε ότι ήταν τόσο υψηλά τα τέλη περιαγωγής που ήταν αδύνατο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν ήταν βιώσιμη. Επίσης, ε, οι πάροχοι υπηρεσιών μας προειδοποιούσαν ότι αν καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής θα οδηγηθούν στη χαροκοπιά. Τελικά, τίποτα αρνητικό δεν έγινε. Ας μην περιμένουμε λοιπόν ε, τόσο πολύ και για μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε τα τέλη της ε, κοινοβουλευτικής μας θητείας για να περιμένουμε το 2018 πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προτάσεις. Ευχαριστώ. Ε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αν ήταν εύκολα θα είχαμε βρει λύση πολύ νωρίτερα. Γιατί το θέμα ε, είναι να βρεθεί μια λύση και να εξορροπηθούν τα διάφορα συμφέροντα. Δεν υπάρχει μόνο Γενική Διεύθυνση Γεωργία, υπάρχουν και άλλε γενικέ διευθύνσει και μερικέ φορέ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί έχουμε τον Επίτροπο Χόγκαν και συμφωνώ ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση και στι υπόλοιπε γενικέ διευθύνσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ο Επίτροπο Χόγκαν είναι με το μέρο μα, αλλά υπάρχουν άλλε διευθύνσει που κολλησιεργούν. Εμεί πάντω συμφωνούμε και συμφωνώ ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Επίση, όπω είπαμε, οι περισσότερε χώρε έχουν α, θεσπίσει και εθνικά μέτρα, αλλά επειδή έχουμε ενιαία εσωτερική αγορά, χρειαζόμαστε πανευρωπαϊκά μέτρα. Ε, μέτρα α, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί έχουμε κάποιε έμεσε ή μάλλον άμεσε πωλήσει, υπάρχουν κάποιοι κάποιες περιπτώσεις για να ε, περιορίσουμε αυτές τις αθεμίτες ε, εμπορικές πρακτικές, ίσως στα βραχιά κυκλώματα διανομής, αλλά δεν αρκούν. Και επίσης έχουμε συγκέντρωση και από μεγάλες πολυεθνικές, αλλά έχουμε και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενεργοποιούνται στον κλάδο. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Θα μπορούσαν να, να συνεργαστούν κάλλιστα και οι συνεταιρισμοί μεταξύ τους. Έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση απέναντι στις αλυσίδες διανομής. Είναι πολύ πιο ενισχυμένη η παραγωγή όταν οργανώνονται σε συνεταιρισμούς ή άλλες οργανώσεις. Επίσης, μερικοί λένε τι να κάνουμε, ε, αυτή είναι η αγορά. Γνωρίζουμε τι χαρακτηριστικά έχει η αγορά και πώς λειτουργεί. Αλλά σίγουρα και οι γεωργοί χρήζουν κάποιες υποστήριξεις και κάποια ρύθμιση είναι απαραίτητη. Δεν μπορούμε να παθαίνουμε μόνο στην αυτορύθμιση. Για παράδειγμα, είδαμε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές α, ε, ε, δεν μπόρεσαν να αυτορυθμιστούν και οδηγηθήκαμε στη χρηματοπιστωτική κρίση που μας ανάγκασε να λάβουμε κάποια υποχρεωτικά ρυθμιστικά μέτρα. Το ίδιο χρειάζεται και εδώ. Να μην τα αφήσουμε όλα στην αυτορύθμιση. Και θα πρέπει στην κοινοβουλευτική μας θητεία και μέχρι το πέρας ε, να καταλήξουμε σε κάποια ευρωπαϊκά νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Γιατί αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο, έγιναν πολλές συζητήσεις, πολλοί άριθμες προτάσεις, θα, περάσουμε, θα πρέπει τώρα να περάσουμε στην επόμενη φάση, στα έργα. Οι δεμοί θα μας κατηγορήσουν οι ψηφοφόροι μας και οι Γεωργοί ότι δεν ανταποκριθήκαμε στο έργο μας και δεν ανταπεξέλθαμε στο ύψος των περιστάσεων, αν δεν καταλήξουμε σε αυτά μέτρα. Ευχαριστώ θερμά τους Υπουργούς για την παρουσία τους, ε, για την παρουσίαση του εγγράφου τους. Φάνηκε από τη συζήτηση πόσο σπουδαίο είναι αυτό το θέμα, αλλά φάνηκε και μία σύμπνοια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να άλληλο βοηθηθούμε και να άλληλο υποστηριχθούμε για να προωθήσουμε αυτό το ζήτημα. Και σίγουρα κάποιες διατάξεις θα ληφθούν υπόψη και στο τριμερή διάλογο για το κανονισμό του Omnibus. Σας ευχαριστώ. Ε, προχωρήσαμε αρκετά, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα πολύ λεπτό τεχνικό διάλειμμα, ένα-δύο λεπτά. Ε, Ξέρω ότι αφιερώσαμε αρκετό χρόνο, αλλά δεν ήθελα να περιορίσω τους καλεσμένους μας λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος. Σε λίγο θα περάσουμε στην έκθεση Μπούντα, ένα-δυο λεπτά, ένα τεχνικό διάλειμμα. Otwieramy wznawiamy obrady, proszę Państwa. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας, ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με ενημέρωσαν ότι ο Υπουργός ε, Γεωργίας Σλοβενίας είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και μάλιστα πρώτος στη τάξη κάτι που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην παρουσίαση αυτού του ανεπίσημου εγγράφου. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το σημείο 5, που προβλέπει την προσαρμογή στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο. Πολύ έξυπνος και περίπλοκος αυτός ο τίτλος της έκθεσης για την οποία αρμόδια κατ' ουσία είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και εμείς θα συντάξουμε γνωμοδότηση που την έχει αναλάβει ο κύριος Μπούντα. Ε, ήδη στην συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου του 2017 αποφασίσαμε να συντάξουμε γνωμοδότηση στην έκθεση Επιτροπής Ιούρη ε, για το, τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο και την ευθυγράμμιση με τα άρθρα 290 και 291. Ο στόχος της πρώτης αυτής είναι η ευθυγράμμιση πολλών νομικών πράξεων που περιλαμβάνουν κάποιες σημείες πριν τη διαδικασία της Λισαβόνας και τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο ε, και προτείνουμε προσαρμογή στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά το νέο καθεστώς για τις ε, καταξιδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Θα μας εξηγήσει τα της διαδικασίας και της ουσίας ο αρμόδιός μας, ο συντάκτης γνωμοδότησης, ο κύριος Μπούντα. Θα μας διαφωτίσει για να καταλάβουμε και να συλλάβουμε σε όλη την περιπλοκότητα το θέμα αυτό. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως θα παρατηρήσατε και εσείς και οι συνάδελφοι, και ο ίδιο ο τίτλος ε, υποδεικνύει πόσο τεχνικό είναι το θέμα αυτό που καλούμαστε να συζητήσουμε. Είναι παρόλα αυτά απαραίτητο. Γιατί στο σημείο αυτό συζητάμε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, την 186 για, την, ε, για τον τερματισμό και την προσαρμογή διαφορετικών πράξεων. ω Επιτροπή Άγκρη Υπάρχουν διάφορε τέτοιε νομικέ πράξει τι οποίε έχουμε εγκρίνει. Είναι σημαντικέ και απαραίτητε αυτέ οι αλλαγέ ε, από τη συνθήκη τη Λισαβόνα και μετά και στο πλαίσιο τη ε, μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική, πολλέ από τι νομοθετικέ πράξει που ακόμα είναι σε ισχύ σήμερα δεν έχουν ακόμα προσαρμοστεί στην ε, νέα διαδικασία συναπόφασης. Καταρχάς, να πω ότι διάβασα την έκθεση Σάιερ του Δεκεμβρίου του 2013 αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά εκτελεστικές αρμοδιότητες. Όπως σας είπα, η διαχωρισμός μεταξύ των εκτελεστικών πράξεων και των πράξεων κατά εξουσιοδότησης είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα, γιατί ουσιαστικά το θέμα είναι τεχνικά ζητήματα. Τεχνικά ζητήματα όπου χρειάζεται να υπάρχει και κάποια αρμοδιότητα στον τομέα, για παράδειγμα, τη Οι τεχνικές αυτές αποφάσεις μπορεί να έχουν και πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ζητά εντολή για πράξεις κατά εξουσιοδότηση, το οποίο θα οδηγούσε σε γενικότερες αρμοδιότητες που θα επηρεάσαν και τον βασικό κανονισμό. Αυτό τι σημαίνει ότι ο κεντρικός ε, κανονισμός θα τροποποιούταν στην περίπτωση αυτή, καθώς και τα προσαρτήματα αυτού. γιατί ό,τι ισχύει για τον κανονισμό ισχύει και για τα παρατήματα και για τα μητρώα και για τις καταλόγους των ε, εγκεκριμένων προϊόντων. Μόνο έτσι μπορεί να μοναγγηθούμε την νομική ασφάλεια. Υπό το φως λοιπόν των προηγούμενων εμπειριών, όπου έχουμε δει πολλά θέματα να μπλοκάρονται και στον τομέα της ε, Επιτροπή Άγκρη και στον τομέα της Επιτροπή Αλία και σε ό,τι αφορά και τα, τον τριμερή διάλογο μετά την πρώτη ανάγνωση. Το Κοινοβούλιο στο σημείο λοιπόν αυτό θα ήθελε να χορηγήσει περαιτέρω τεχνικές αρμοδιότητες προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη αρμοδιότητα για την προστασία του καταναλωτή. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τη συντροποποίηση 768 νομοθετικών πράξεων, αλλά η πιο σημαντική εξ αυτών είναι ο κανονισμός 767 του 2009. Αυτό σημαίνει η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα ασχοληθεί με τον κανονισμό αυτό και όχι με άλλους που δεν ε, από τον άμεσα του γεωργικού κλάδου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο, το άρθρο 290 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ σε κάποια σημεία ορίζεται υπό ποιους όρους μπορεί να ισχύσει το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις οτροφές. Επίσης, ό,τι αφορά τον κατάλογο για τα χημικά με ανώτατες περιοκτικότητες σε κάποιες ουσίες. Επίσης, ε, να σας πω ότι οι αρμοδιότητες αυτές για τις πράξεις κατά δεν χορηγούνται εφάπαξ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο για περίπου 5 ετών. Και έτσι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν στις αρμοδιότητες αυτές. Μετά από 9 μήνες λοιπόν ανάθεση της αρμοδιότητας ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να καταθέσει έκθεση για παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης. Ε, φυσικά, αυτό επηρεάζει πολλές νομοθετικές πράξεις, αλλά μόνο αυτές οι δύο που σας ανέφερα είναι σημαντικές για εμάς ως Επιτροπή Γεωργίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καπούτο είναι ο πρώτος μας ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Παουλούτσι είναι ο σκιώδης εισηγητής για το σημείο αυτό και εκφράζει εκ μέρους των σοσιαλιστών. Όμως δεν μπόρεσε να έρθει το Βρυξέλλες και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπούντα για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, συμφωνούμε με αυτό. Ε, κάποιες περιπτώσεις φακέλων που αφορούν την ευθυγράμμιση των νομοθετικών πράξεων ε, είναι ουσιαστική ε, για τη γεωργία. Ε, και πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά την κατάρρευση των τριμερών ε, διαλόγων της πρώτης ανάγνωσης. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα τεχνικά θέματα που να επηρεάσουν τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Όμως, είναι σημαντικό η υιοθέτηση κατεξουσιοδότηση πράξεων να είναι μια αρμοδιότητα που θα δίδεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πέντε χρόνια ανεώσιμα, ε, όχι όμως επαορίστο, όπως θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να αφορά όλες τις, ε, τα κείμενα της ε, Επιτροπής Άγκρη, καταρχάς ας πούμε για τις ζώοτροφές, όπως παραδείγματος τα κείμενα για τις ζωοτροφές, κάποιες ζωονόσους κτλ. Ε, θα υποβάλει ο κ. Παουλούτσι κάποιες τροπολογίες προς, ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να δουλέψει ε, με θετικό πνεύμα. Ε, και πιστεύω ότι αυτές οι τροπολογίες ε, γενικά θα βρουν σύμφωνους ε, τους σκιώδες και ένα μεγάλο μέρος των Ευρωβουλευτών της Επιτροπής. Ο κ. Στάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της, του Άλντε, ευχαριστώ τον κύριο Μπούντα. Καλό και ισορροπημένο το σχέδιο της νομοδότησής του. Η ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ δύσκολη. Τσίμα-τσίμα πέρασαν κάποια πράγματα. Η κατεξιοδότηση πράξης είναι ένα πολύ λεπτό πολιτικό θέμα. Γι' αυτό ακριβώς Πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά αυτή την πρόταση στην Επιτροπή Γεωργίας. Είναι σημαντικό να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία. Αφορά τις νομοθετικές μας πράξεις. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τις κατεξιοδότηση πράξης και για την μεταβίβαση ε, εξουσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υιοθετεί τέτοιε πράξεις. Ειδικά σε κάποιους τεχνικούς τομείς είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε τους ε, ειδικού που συντάσσουν τις προτάσεις και είναι σημαντικό αυτοί οι εμπειρογνώμονε να προέρχονται από τα κράτη-μέλη και τι ομάδες συμφερόντων. Ε, μία ερώτηση προ τον κύριο Μπούντα. Γιατί θέλουμε ορισμούς ε, τους ορισμού μάλλον των ζωοτροφών να αποφασίζονται μέσω καταξιωτότηση πράξεων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μπορώ να κάνω αυτή την ερώτηση προ τον κύριο Μπούντα. Δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο από την Ομιγύρη. Οπότε θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπούντα, για να απαντήσει. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε σίγουρα να συζητήσουμε το γιατί θα πρέπει να οριστεί ο όρος ζωοτροφές, μιας και υπάρχει ίδιο ορισμός, αλλά... Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και μια συζήτηση στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την τροποποίηση διάφορων νομοθετικών πράξεων. Πώς λοιπόν μπορούν αυτές οι αλλαγές να επέλθουν για τα τροφήμα για τις ζωοτροφές, για τα φάρμακα, γιατί στην αγορά, ξέρετε, υπάρχουν εξελίξεις. Αυτό που σήμερα ορίζεται ως τροφή μπορεί σε πέντε χρόνια να χρήσει νέου ορισμού. Το ερώτημα είναι το πώς θα γίνει αυτή Πώς θα καθοριστεί ο νέος ορισμός, θα γίνει μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω πράξεων κατά εξουσιοδότηση ή θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό ακριβώς, κατά πόσο θα συμμετάσχει το Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή. Και γι' αυτό λοιπόν προτιμώ τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, προκειμένου να έχει λόγο και το Κοινοβούλιο. δεν πιστεύω ότι έχει ζωφερούς σκοπούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα αυτά μόνο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποιους τομείς όπου ο καιρός έχει και η εμπειρία έχει καταδείξει ότι ενδεχομένως να μην έχει τις απαραίτητες πληροφορίες στη διάθεσή της. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. προκειμένου να μπορούμε στη συνέχεια να παρουσιάσουμε στη δημόσια γνώμη μια ενημερωμένη, ενημερωμένο έγγραφο. Έχετε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 26 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι. Αν δεν υπάρχουν άλλες απορίες, ε, παρατηρήσεις, σχόλια, μπορούμε να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες και τα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης. ευχαριστώ. Καλό βράδυ.